Καλημέρα αγαπητοί συνάδελφοι. Αρχίζουμε λοιπόν την συνεδρίαση της Επιτροπής μας και πρώτα απ' όλα να την ημερήσια διάταξη. Αν δεν θέλετε καμία αλλαγή, τότε θεωρείται και εγκεκριμένη. Δεύτερο σημείο, ανακοινώσει της Προέδρου. Έχουμε τη Σίλα Βέρικα από το ECR που ήρθε στην Επιτροπή μας ως αναπληρωματικό μέλος. Σήμερα είναι μια πολύ σημαντική μέρα για την Πορτογαλία και για τις γυναίκες. Για το ζώο Πιμέντα, ο αντιπρόεδρος μας, ναι. έχει γενέθλια σήμερα. Αγαπητοί συνάδελφοι, πάμε στο επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη τώρα που είναι η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Έχετε τις κάρτες σας, σωστά. Οπότε αρχίζουμε και την ψηφοφορία. για μια εξωτερική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση των πρόωρων γάμων. Επόμενα βήματα. Είναι γνωμοδότηση και συντάκτρια της γνωμοδότησης αυτής είναι η Ντανιέλα Γιούτο. Συμβιβαστική 8. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 45. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 46 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 52, σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 48, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 9 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 54 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 10 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 51 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 11 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 63 υπέρ, κατά, αποχές. Θα ελέγξουμε εδώ για την τροπολογία 63 παρακαλώ. Μπορείτε να ψηφίσετε. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συγγνώμη που σα έβαλα να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά, να σηκώνετε όμως τα χέρια για να σας βλέπω, γιατί αλλιώ δεν ξέρω. Τροπολογία 91 τώρα, σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Να ελέγξουμε, ωραία, να ελέγξουμε. 91 δεύτερο τμήμα. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 89 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 71 κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 78. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 69. Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται νομίζω, αλλά θα ελέγξουμε καλύτερα για την τροπολογία 69. Πρώτο τμήμα ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε. Τέλος της ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. 69. Όχι, το δεύτερο τμήμα δεν το ψηφίζουμε. Ωραία, πάμε στην τροπολογία 70 τώρα. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 72 υπέρ. Κατά αποχές, εγκρίνεται. 73 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 13 τώρα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 14 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 97 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 79 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 80 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 15 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 76 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 77 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 16 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 81 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 95 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 55 με προφορική τροποποίηση υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 90 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 93 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 94 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται.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 κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 87 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 100 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 47 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 101 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 82 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τώρα πάμε σε τη σκέψη. συμβαστική αριθμός 1 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 4 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 23 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 6 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 24 υπέρ, κατά, αποχές, Εγκρίνεται. Τροπολογία 36 με προφορική τροποποίηση υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 8 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 17 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 13 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 18 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 33 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 34 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 7 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 15 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 16 υπέρ, κατά, αποχές,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 κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 41 τώρα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα με ηλεκτρονική ψηφοφορία το τροποποιημένο σχέδιο γνωμοδότησης. Μπορείτε να ψηφίσετε παρακαλώ. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Συγχαρητήρια κυρία Αγίουτο και όλους και όλους συζητητές. Σας ευχαριστώ. Προχωράμε. Πάμε στην επόμενη ψηφοφορία. Uh, next vote is ε, monitoring the application of... Παρακολουθώντας την εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου ως αφορά το 2016 έγκριση σχεδίου γνωμοδοτήσεως. Η Μαριάννα Πετήρ είναι η συγχύτρια για τη γνωμοδότηση. Ξεκινάμε. Τροπολογία 33 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 34 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 36 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 42 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 43 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 45 υπέρ κατά αποχές πρέπει να κάνουμε έλεγχο για την τροπολογία 45 άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικός έλεγχος πέρας εγκρίνεται τροπολογία 46 υπέρ κατά Άλλη μια φορά. Υπέρ. Τη 46 παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Έλεγχος. Για τη 46 ξεκινάει η ψηφοφορία τώρα. Πέρας. Εγκρίνεται. Σαράντα υπέρ κατά Άποχες εγκρίνεται. 48 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 50 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 51 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 52 υπέρ κατά αποχές πρέπει να ελέγξουμε την τροπολογία 52 ηλεκτρονικός έλεγχος. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 53 υπέρ. Κατά αποχές έλεγχος για την 53. Άρχεται του ηλεκτρονικός έλεγχος. Πέρας αυτού. εγκρίνεται. Τροπολογία 54 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 56 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Έλεγχος για την 56. Ηλεκτρονικός έλεγχος που ξεκινάει τώρα. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 9 υπέρ. Υπέρ παρακαλώ, τροπολογία 9. Κατά. Άποχες. Έλεγχος σας παρακαλώ. Τροπολογία 9, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 1 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 12 τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 14 σε τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα υπέρ κατά αποχές έλεγχος για το τρίτο τμήμα σας παρακαλώ, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Απορρίπτεται. 15 υπέρ. Κατά αποχές έλεγχος για την τροπολογία 15 που ξεκινάει τώρα. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τοπολογία 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Έλεγχος. τοπολογία 18 άρχεται ο ηλεκτρονικός έλεγχος. Πέρας. Εγκρίνεται. τοπολογία 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 22 σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 24 σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ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 εγκρίνεται. Τροπολογία 31 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 32 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία. Θέλετε να κάνουμε παλήθευση για 32. Καλώς. Ηλεκτρονικός έλεγχος για 32. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται, εγκρίνεται. Πάμε στην τροπολογία 1 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Να ψηφίσουμε μαζί τη 2 και την 8 ή όχι. Να ψηφίσουμε μαζί. Ναι. Τροπολογία 2 μέχρι την 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Πάμε ηλεκτρονικά το σχέδιο γνωμοδοτήσεως που τροποποιήθηκε, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας εγκρίνεται. Συγχαρητήρια λοιπόν στην εισηγήτρια Μαριάννα Πετήρ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε στην επόμενη ψηφοφορία. Σημείο 5 στην ημερήσια διάταξη. Παραβίαση των δικαιωμάτων των ηθαγενών πληθυσμών ε, στην, ε, στον κόσμο και αρπαγή γεών, υιοθέτηση σχεδίου γνωμοδοτήσεω. Φλόρεν Μασελεύσιφ. Εισηγητής. Είσαστε έτοιμοι για ψηφοφορία. Συμβιβαστική ένα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 15 υπέρ, 15 υπέρ παρακαλώ κατά αποχές εγκρίνεται 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 17 υπέρ κατά αποχές πρέπει να γίνει επαλήθευση για τροπολογία 17 άρχεται η ψηφοφορία Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 18 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 19 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 20 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 21 υπέρ. Κατά αποχές θα κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο για τροπολογία 21 ξεκινάει η ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται τροπολογία 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τροπολογία 29 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 30 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 36 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 37 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 38 υπέρ κατά αποχές. Παρακαλώ να κάνουμε έλεγχο η τροπολογία 38. Άρχεται η ψηφοφορία. 38. Ξεκινάμε. Τέλος. Απορρίπτεται. Τροπολογία 39 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 40 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 6 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Θέλετε να ελέγξουμε τη συμβιβαστική 4. Έλεγχος λοιπόν για τη συμβιβαστική 4. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 47 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 48 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 49 λέει πρόεδρος, πρώτο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, τη 49 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 50 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 51 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 52 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 53 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 55 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 56 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 57 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 58 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 59 υπέρ έλεγχος. Θέλετε έλεγχο για την 58. Άρχεται η ψηφορία για την τροπολογία 58. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 59 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας ελέγξουμε την 59. Άρχεται ηλεκτρονικός έλεγχος. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 60 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 1 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ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 κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και τροπολογία 10 υπέρ υπέρ παρακαλώ κατά αποχές εγκρίνεται. και θα ψηφίσουμε το σχέδιο γνωμοδοτήσεως που τροποποιήσαμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται και συγχαρητήρια στον συνάδελφο Φλωρένς Μασελέση. Ευχαριστώ πολύ. It was the end of Ολοκληρώσαμε λοιπόν τι ψηφοφορίε. Μπορούμε να περάσουμε στα διάφορα, αν υπάρχει κάτι. Και θέλω να σα ενημερώσω ότι η επόμενη συνεδρίασή μα θα πραγματοποιηθεί στι 25 Απριλίου το πρωί από τις 9 έως τη 1 το μεσημέρι. Uh, uh, uh, Επόμενο σημείο της σημερινής διάταξης είναι το δίκτυο για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου και η συζήτηση για το θέμα αυτό θα ξεκινήσει στις 10. Τώρα διάλειμμα και επανερχόμαστε στις 10.